Welcome to everybody. We can start our meeting, you know. Καλώς ήρθατε όλοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ξέρετε ότι η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και θα μιλήσω Ιταλικά στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης και μετά στα Αγγλικά ξανά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια σημαντική υποχρέωση που πρέπει να φέρουμε εις όπως και πολλές άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πρέπει να ορίσουμε, να εκλέψουμε την νέα επίσημη το νέο επίσημο πρόεδρο. Ο συνήθως είναι web stream τη συνεδρίασή μα και βάσει το άρθρο 204 για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των υπόλοιπων Αντιπροέδρων θα κάνουμε εδώ όσα προβλέπονται και μετά τις εκλογές την, ε, τα, ε, τη σκητάλη θα την, παραδώσω στον ε, νέο εκλεγέντα ή την νέο εκλεγήσα πρόεδρο. Θα έλεγα να περάσουμε αμέσω στην ψηφοφορία. Δεν έχω αποβάλει εγώ ίδια την υποψηφιότητά μου, διότι υπήρξε συμφωνία εντό των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην αρχή τη θητεία και είχαμε αποφασίσει για τα μισά αυτή να υπάρξει εναλλαγή. Να πω λοιπόν ότι για μένα αυτή η εμπειρία των 2,5 αυτών ετών ήταν πλούσια και ιδιαίτερα πρόσφορη και σας ευχαριστώ όλους για την στήριξη, την κατανόηση και τη γενναιοδορία με την οποία συνεργαστήκατε μαζί μου ως ε, ένα σώμα σε, τόσο, σε πολλά δύσκολα εγχειρήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και όλος ιδιαιτέρως τους και τις αντιπροέδρους. Τέσσερις αυτοί. Τρούπελ, Μπόξερ, Διακόνου και τους συντονιστές των ομάδων και της δικής μου ομάδας και βεβαίως όλους τους συναδέλφους ε, βουλευτές τους ε, συνεργάτες μας, ε, τους βοηθούς και την ίδια τη γραμματεία για την πολύτιμη προσφορά της και την πιστή παρουσία της και αφοσίωσή της. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για την πολύτιμη βοήθειά σας. Πριν ξεκινήσω, νομίζω πρέπει να θυμίσω και με συγχωρείτε αυτήν την τραγωδία που συνέβη στη χώρα μου σε δύο διαφορετικά ε, περιστατικά. Πρώτα απ' όλα με το λεωφορείο με τους 16 Ούγγρους φοιτητές, οι οποίοι έχασαν τη ζωή, της, τη ζωή τους. Φανταστείτε ότι επέζησαν κάποιοι από τους γονείς και τους δασκάλους, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι νεότεροι που καθόντουσαν πίσω. Είναι μια τραγική στιγμή που χτυπάει το άνθος της νιώτης στην Ευρώπη και αυτό πραγματικά είναι κάτι που αξίζει να το αναφέρουμε και ακόμη όσους είναι χαμένοι ακόμα ε, κάτω από το χιόνι στο Αμπρούτσο ε, με τον ε, σεισμό και την χιονοστιβάδα που ακολούθησε. Θα σας ζητήσω λοιπόν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα αυτών των τραγωδιών. Πάντα προέχουν οι άνθρωποι και μετά θα περάσουμε στην πολιτική μας υποχρέωση. Grazie. Bene. Ωραία. Και τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη, και του Πρόεδρου. Προηγουμένως, να σας ενημερώσω τι αναπληρωτέ έχουν προταθεί από τους ομάδε ΕΛΚ. ΕΡΝΤΟΚ. Που δικαθιστά τον κύριο Ζαγοράκη. Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε Σίλβια Κάουφμαν. Στη θέση του κύριου Γραμματικάκη. Ιβαν Κάταλιν Σόριν. Αντί για τον κύριο Ντράγκητσι. Άλντε Σφόρ. Γοσφό. Για τους πράσινους ο, Ραμόν, ο κύριος Ραμόν στη θέση τη κυρία Εύαν, συντηρητικούς και, μεταρρυθμιστέ συντηρητικοί μεταρρυθμιστέ μεταρρυθμιστές Γιαννοντεύσκη, στη θέση ποιου δεν υπάρχει εδώ το όνομα, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιος αντικαθίσταται. Μπορείτε να μα το πείτε. Για του συντονιστέ λέτε. Χρειαζόμαστε μόνο το όνομα αυτού που αντικαθίσταται. Μπορείτε να ρωτήσετε τη σύμβουλό μου. Τέλεια. Άλλες αντικαταστάσεις που πρέπει να ανακοινώσω. Ωραία. Εάν υπάρχει κάτι άλλο, πείτε μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει απαρτία 8 μελών, 1 ε, τέταρτο των μελών και Τώρα η ανακοίνωση της υποψηφιότητας για την Προεδρία. Να δώσω το λόγο στο μέλος που θέλει να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του. Πρώτα απ' όλα κυρία Λιμπάτσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προτού παρουσιάζω την υποψηφιότητα της κυρίας Πέτρα Κάμερεβερτ, ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω εσάς για το έργο σας, κυρία Πρόεδρε. Ήταν μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε. Και τώρα, και πάλι, είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ να σας παρουσιάσω την υποψηφιότητα της κυρίας Πέτρα Κάμερεβερτ. Η συνάδελφός μας είναι εξαιρετικά ε, ικανή δραστήρια στους σοσιαλιστές και δημοκράτες και έχει εργαστεί ανέκαθεν πολύ σκληρά. Ε, ανέκαθεν ήταν άκρος επαγγελματίας στην ε, στάση της, ότι αφορούσε τα μεμονωμένα ντοσχέ, τα οποία αναλάμβανε ως εισηγήτρια. Είμαι βέβαιη ότι με την προεδρία τη συναδέλφου Κάμερε Βέρτη, η Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευση θα λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά, πρόσφορα και ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε αρμονικά και με τους βουλευτές άλλων επιτροπών και τους αρμόδιους επιτρόπους. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να στηρίξω την υποψηφιότητα αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε Κριστίνα. Καταγράφουμε την υποβολή αυτής της υποψηφιότητας. Ρωτώ βάζει και του κανονισμού αν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι, άρα Περνώ ευθύ αμέσω. Πρέπει καταρχάς να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία Μπράβο σας κυρία Καμερέφερτ. Ε, τα στοιχεία που επιτρέπουν να υποβάλει υποψηφιότητα η κυρία Καμερέφερτ, ότι είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής Κάλτ, ότι εκπροσωπεί μια πολιτική ομάδα και έχει υποβάλει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει καμία συμβατότητα. Οπότε, θα ζητήσω από την ίδια την υποψήφια, την κυρία Πέτρα Κάμερεβερτ, να μας πει αν δέχεται την υποψηφιότητα και αν θέλει να αναλάβει ως πρόεδρος. Ναι, Άρα, θερμές ευχές, συγχαρητήρια κυρία Κάμερεβερτ. Και επειδή δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, θα έλεγα να κηρύξουμε εκλεγμένη την κυρία Καμερέβερτ. Διαβόησε, έτσι, δηλαδή, εφόσον όλοι συμφωνούμε, έχει εκλεγεί. Συγχαρητήρια κυρία Καμερέβερτ και συγχαρητήρια Πέτρα. Ωραία. Προ στιγμή η δική μου υποχρέωση, από αυτή τη μεριά τουλάχιστον του Προεδρείου, έχει ολοκληρωθεί. Πέτρα, σε καλό να αναλάβει την Προεδρία τη Επιτροπή με μεγάλη χαρά και μετά θα περάσουμε στην εκλογή των τεσσάρων αντιπρόεδρων. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους. Πέτρα. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας καταρχάς. Δεν θέλω να αρχίσω όμως τη δουλειά μου χωρίς να ευχαριστήσω ότι μέχρι τώρα ε, πρόεδρό μας, την κυρία Σίλβια Κώστα, για την εξαιρετική πραγματικά και καταπληκτική της δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίλβια, αυτά είναι πολύ ειλικρινά που λέω και από την καρδιά μου. Δυόμιση χρόνια έκανες πολύ σκληρή δουλειά εδώ στην Επιτροπή, πραγματικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήγες μπροστά την Επιτροπή Πολιτισμού, αύξησε την προβολή της και την ε, εικόνα της. Ελπίζω να μπορέσω να συνεχίσω στο δρόμο που χάραξες εσύ και να διαμορφώσω κι εγώ λίγο το μέλλον για την Επιτροπή μας. Και προσβλέπω σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, καλή συνέχεια και ευχαριστώ πολύ.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 λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπό μου. Ελπίζω και θα αγωνίζομαι κάθε στιγμή γι' αυτό να είμαι δίκαιη πρόεδρος και ε, θα συνεχίσω στη γραμμή που χάραξε η Σίλβια Κώστα και θα κάνω ό,τι μπορώ για να ε, προβάλλω και να εκπροσωπώ ε, την Επιτροπή Πολιτισμού όχι μόνο προς τα έξω αλλά και στο εσωτερικό να φροντίζουν να έχουμε ένα καλό κλίμα εργασίας και μια ατμόσφαιρα έτσι ώστε ε, να καταλάβουν και άλλες επιτροπές που καμιά φορά δυσκολεύονται ότι η Επιτροπή Πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικά ε, θέματα να διεκπεραιώνει και να μην χάνεται. Ε, πραγματικά πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια αυτή η Σιλβία Κώστα και ελπίζω να το συνεχίσω κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε και άλλες εκλογές τώρα, μερικές ε, ε, Άντρες και γυναίκες. Έρχομαι μέσα στην εκλογή της πρώτης αντιπροέδρου και πάλι για λόγους τάξεως και ε, τύπου θα πρέπει να σας πω ποιοι είναι παρόντες σήμερα και ποιοι προτείνονται. Μάλλον ποιος εκπροσωπεί τον κύριο Ζαγοράκη, ο συνάδελφος ε, ε, Νόρμπερτ Έρερς, ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η κυρία Κάουφμαν έχει έρθει στη θέση του κύριου Γραμματικάκη. Ο Καταλήν Σόρεν Ήβαν εκπροσωπεί τον συνάδελφο και από την Άλντε ο Ρόμπερτ Χωσφό, εκπροσωπεί τη συνάδελφο Γιάννα Τόμ. Και από τους Πρασίνους, ο κύριος Ραϊμόν ε, εκπροσωπεί ε, τη συνάδελφο που απουσιάζει και το ECR, ο συνάδελφος Μέσσερ Σμιτ απουσιάζει και τον αντικαθιστά κύριο Κρασοντεύσκη. Άρα, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε 8 μέλη τουλάχιστον για να εξασφαλίσουμε την απαρτία. Και παρακαλώ υποψηφιότητε. Η Σαμπίνα Φερχάιν. Θα ήθελα καταρχά και εγώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τη Σίλβια Κώστα για την εξαιρετική δουλειά τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Ήταν πάρα πολύ ειλικρινή η συνεργασία μα και πάρα πολύ άξια εκπροσώπησε ε, την Επιτροπή μα. Θέλω να τη ευχηθώ ότι καλύτερο για τη μελλοντική της ε, εργασία και καλή συνεργασία εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών εκείνη. Και εσύ, Πέτρα, ότι επιθυμείς καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα και ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε την καλή συνεργασία που έχουμε. Είναι σε καλά χέρια η Επιτροπή μας και μετά από αυτή την αλλαγή φρουράς. Έχουμε σημαντικά θέματα, το είπες και εσύ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα που δεν αναγνωρίζουν πάντα όλοι, ούτε μα παίρνουν όλοι στα σοβαρά εδώ, οι άλλε επιτροπέ δηλαδή του Κοινοβουλίου. Άρα θα πρέπει να διατρανώσουμε ότι ο ρόλο ε, τη επιτροπή μα είναι σημαντικό. Θέλω να προτείνω την κυρία Ανδρέα ε, Μπόξορ από ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ω πρώτη αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ. άλλε προτάσει υπάρχουν? Όχι, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, η κυρία Ανδρέα Βόξχορ είναι πλήρες τακτικό μέλος ε, της Επιτροπής μας, προτείνεται από μια πολιτική ομάδα, έχει καταθέσει και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων της, οπότε ε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για την εκλογή της. Θέλω να τη ρωτήσω και επίσημα αν αποδέχεται ε, την υποβολή της υποψηφιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, την αποδέχομαι μια που είναι η μοναδική υποψήφια θα πρότεινα να την εκλέξουμε διαβοής. Θέλει κανείς να γίνει μυστική ψηφοφορία. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Να την εκλέξουμε λοιπόν δια βοής παρακαλώ την κυρία Πόσκο. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε. Σας παρακαλώ να έρθετε εδώ να καθίσετε στο πλευρό μου. Μετά, Εφτάσαμε ήδη στο δεύτερο αντιπρόεδρο και εδώ πάλι για λόγους τύπους θα πρέπει να ε, εκφωνήσω τα ονόματα των βουλευτών που αντικαθιστούν κάποιους συναδέλφους για το ΕΛΚ. Αποουσιάζει ο κύριος Αγοράκης, τον οποίο αντικαθιστά ο κύριος Νόμπερτ Έζερς. Τον κύριο Γραμματικά και από τους σοσιαλιστές ε, αντικαθιστά η κυρία Κάουφμαν ε, και για τις άλλες πολιτικές ομάδες Ντράγκη Σόριν για έναν Τόμ στην Άλντε εκπροσωπεί ο κύριος Ροσφόρ. Ε, Εύαν των Πρασίνων απουσιάζει και είναι στη θέση του Ρεμόν και ο κύριος ε, Κρασνοντεύσκη είναι στη θέση του κυρίου Μέσσερ Σμιτ. Έχουμε αρκετό αριθμό μελών που παρευρίσκονται, 8 χρειάζονται για την απαρτία και είμαστε πολύ περισσότεροι Πρόταση λοιπόν για τη θέση του Δευτέρου Αντιπροέδρου. Παρακαλώ. Καταρχάς, συγχαρητήρια ε, Πέτρα για την εκλογή σου. Θέλω να πω στη Σίλβια ότι ήταν σπουδαία πρόεδρος και ε, θα μας λείψει. Η ομάδα μας προτείνει τον κύριο Μιρτσέα Διακόνου να συνεχίσει να παρέχει τις καλές υπηρεσίες του που όλοι γνωρίζουμε. Έχει διαταλέσει αντιπρόεδρος και η ομάδα των φιλελευθέρων τον προτείνει ως δεύτερο αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλες υποψηφιότητες, άλλες προτάσεις. Όχι, δεν βλέπω. Οπότε διαπιστώνω ότι ο κύριος Διακόνο είναι Πρώτον, τακτικό μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού. Δεύτερον, προτείνεται από μια πολιτική ομάδα. Και τρίτον, έχει υποβάλει τη δήλωση οικονομικών του συμφερόντων. Και πάλι, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για να τέθει η υποψηφιότητά του σε ψηφοφορία. Συμφωνείτε με την υποψηφιότητα αυτή, κύριε Διακόνο. Ναι. Μάλιστα, αλλά θα προτιμούσα κάποιος ε, άλλος να είναι σε θέση να οριστικοποιήσει τον τριμερή διάλογο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς νομίζω θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, διαπιστώνω ότι ε, είναι ένας και μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Δευτέρου Πρόεδρου και θα πρότεινα και εδώ να εκλέξουμε διαβοή του συνάδελφου Διακόνου. Δεν έχει ζητήσει κανείς μυστική ψηφοφορία. Ωραία. Προχωρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Θερμά. Και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία μαζί σας και χαίρομαι γι' αυτό. Σας παρακαλώ ελάτε να καθίσετε στο Προεδρείο τρίτος αντιπρόεδρος ή τρίτη αντιπρόεδρος. Το αυτό ως διαδικασία. Πάλι πρέπει να σας αναγνώσω τα απόντα μέλη και πιο στους εκπροσωπεί Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Λείπει ο κύριος Ζαγοράκης. Τον αντικαθιστά ο κύριος Νόρμπερτ Έρδερς. Ε, Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Η κυρία Κάφμαν καθιστά τον κύριο Γραμματικάκη. Δάμια Γκραγκίξη ε, ε, λείπει και ο Σορή. Γομπέ ε, από τους Φελελευθέρους και ο κύριος Ραϊμόν αντικαθιστά την κυρία Εύανς και ο κύριος Κραζοντέψ και τον κύριο Ροσφό, τον κύριο Μέσα Σμίτ, συγγνώμη. Ε, προτάσεις. Ο κύριος Ραϊμόν. Ευχαριστώ. Καταρχάς, εξ ονόματος των Πρασίνων, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τη Σίλβια Κώστα ε, για τη διεύθυνση της Επιτροπής μας όλα αυτά τα χρόνια και να συγχαρώ την πρόεδρό μας και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί. ε, πορεία αυτή προτείνω τη Χέλγα Τρούπελ για την τρίτη αντιπροεδρία. και δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις, ε, ε, είναι γνωστή και θα εξακολουθήσει να ασκεί τα καθηκοντά της με τον ίδιο τρόπο φανταζόμαι. Άλλες υποψηφιότητες υπάρχουν, όχι και η κυρία Τρούπελ είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής μας. Ε, την προτείνει μια πολιτική ομάδα και έχει υποβάλει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων της. Δεν υπάρχει εμπόδιο για την εκλογή της, δεν υπάρχει ανθυποψήφιος και προτείνω να την εκλέξουμε δύο Α, όχι, όχι, πρέπει να σας ρωτήσω. Να ρωτήσω τη Χέλγα, συμφωνείς εσύ με την υποψηφιότητα. Καλά που το σκέφτηκες. Ναι, ε, καλώς είναι σου. Συμφωνώ, βεβαίως. Ναι, το υπέθεσα, γι' αυτό δεν σε ρώτησα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μία υποψήφια, δεν υπάρχει αντιποψήφιος και προτείνω να την εκλέξουμε διαβοής, αν δεν θέλει κανείς μυστική ψηφοφόρια που δεν θέλει, από ό,τι βλέπω. Auch dir, Helga, ε, συγχαρητήρια, Χέλγα. Ε, ε με βέβαια ότι θα συνεχιστεί η καλή συνεργασία, αλλά και εσύ εδώ στο Προεδρείο. Λοιπόν, και φτάσαμε ήδη στον τέταρτο αντιπρόεδρο. Και πάλι, για τελευταία φορά θα σας πω ποιοι είναι απόντες και από ποιους αντικαθίστανται. Λοιπόν, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κύριο Έρδε, αντικαθιστά τον κύριο Ζαγοράκη. Η κυρία Κάουφμαν από σοσιαλιστέ, τον κύριο Γραμματικάκη. Ο κύριος Καταλήνη Σορινίβαν, τον κύριο Ντράγκινση. του φιλελεύθερου, ο κύριο Ροσφόρ, ε, κάποιον από τα συνάδελφο ε, και τους πρασίνους λείπει η κυρία Εύαν και είναι ο κύριο Ραϊμόν και ο κύριος Κράσνοντεύσκη αντικαθιστά τον κύριο Μέσερ Σμιτ. Προτάσεις παρακαλώ για τον ή την τέταρτη αντιπρόεδρο η Σαμπίνε Φερχάεν. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα ήθελα να προτείνω τον Στέφανο Μάολου ως τέταρτο αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ρωτήσω και τον κύριο Μάουλο αν συμφωνεί με την υποψηφιότητά του. Ναι, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Άλλος, άλλες προτάσεις δηλαδή έχουμε. Όχι. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο και πάλι διότι ο κύριος Μάουλου είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής μας, προτείνεται από μια πολιτική ομάδα και έχει υποβάλει τη δήλωση οικονομικών του συμφερόντων. Και μια που δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, ούτε εδώ, προτείνω να τον εκλέξουμε και εκείνον διαβοή. Αν κάποιο επιθυμεί μυστική ψηφοφορία πρέπει να γίνει, όχι από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, και πάλι εκλέγουμε τον κύριο Μάουλου διαβοή. Συγχαρητήρια θερμά για την εκλογή σα και χαίρομαι και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία και σα παρακαλώ να έρθετε στο Προεδρείο να καταλάβετε τη θέση σα. Νομίζω εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο τμήμα, το επίσημο και το τυπικό και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ μάλλον και μπορούμε να προχωρήσουμε στην κανονική μας συνεδρίαση και στην ημερήσια διάταξη. Πάμε λοιπόν στο σημείο 3 κανονικά. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε επιθυμίες για αλλαγή στην ημερήσια διάταξη? Όχι. Αντιρρήσεις? Όχι. Άρα θεωρείται εγκεκριμένη μέρη σε διάταξη με τη μορφή που σας έχει υποβληθεί το σχέδιό της. Σημείων 4 στη μέση διάταξη. Τα πρακτικά της συνεδρίασης 10-11 ε, Οκτωβρίου, της 8 Νοεμβρίου και της 28 Νοεμβρίου 2016. Τα σχέδια των πρακτικών σας έχουν διανεμηθεί των τριών αυτών συνεδριάσαν. Έχετε παρατηρήσεις για τα πρακτικά αυτά? Όχι. Και προτείνω να ακολουθήσουμε τη συνήθεια διαδικασία. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Φτάσαμε ήδη στο σημείο 5, ανακοινώσεις Προέδρου. έχω να σας ανακοινώσω ότι σήμερα έχουμε διερμηνία στα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, εστονικά, ουγγρικά, πολωνικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Αύριο το απόγευμα θα έχουμε και σλοβενικά. Έχετε επίση τι αποφάσει τη συνεδρία των συντονιστών τη 5η Δεκεμβρίου 2016. Τις ε, λάβατε με mail στις 8 Δεκεμβρίου. Και έχουν εγκριθεί γιατί δεν διαφώνησε κανείς μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου που έληξε η προθεσμία για το σκοπό αυτό. Καλά, υπερταχεία. Δεν έχει έρθει ο εισηγητής για το σημείο 6. Ο κύριος Φίσας. Τώρα έχουμε τις εξή δύο δυνατότητες. Είτε θα εξετάσουμε πρώτα το σημείο 7, που είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο και μια δυνατότητα, και όταν έρθει ο κύριος Φίσας να επανέλθουμε στο 6. Τζούλη. Συγγνώμη για τα πρακτικά. Μόλις παρατήρησα ότι έχει γραφτεί λάθος το όνομα του Ken Loach στη σελίδα 2. Πρέπει να το γράψουμε σωστά, έτσι, με τη σωστή ορθογραφία. Μάλιστα, θα το διορθώσουμε. Θα επιληφθεί η γραμματεία. Δεν είναι δυνατόν να γράφουμε λάθος τα ονόματα. Okay. Ε, Ζαμπίνε. Ζαμπίνε Φεχέν, τι γίνεται με τον Σαντιάγο, θα μας έρθει. Έμαθα ότι δεν θα έρθει. Μόλις τώρα μου το λένε. Και έχω ένα σύντομο σημείωμα για το ίδιο το κείμενο. Δεν ξέρω. Να σας διαβάσω. Α, αν δεν έρθει καθόλου σήμερα, τότε μπορούμε να διακπεράσουμε το θέμα αυτό με το σημείωμα και με διάφορες παρατηρήσεις και τοποθετήσεις των σχεδόν εισηγητών. Απουσία του κύριου Θα μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομη, διότι λέει. Το σχέδιο έκθεση ε, δεν αλλάζει ουσιαστικά την πρόταση τη Επιτροπή. Μοναδικό σκοπό τη έκθεση είναι να, εισαχθούν, ε, να συμπεριληφθούν οι χώρε ΕΦΤΑ και να τροποποιηθεί αναλόγω και το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται. Έχουμε τροποποιήσει μόνο μερικέ παραγράφου για να διευκρινιστεί η έκθεση, αλλά όχι επί του περιεχομένου. Γιατί θεωρούμε ότι ήταν καλή πρόταση ω είχε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ έχει κάνει καλή προεργασία, οπότε δεν άλλαξε ουσιαστικά τίποτα, εκτός από τη διεύρυνση και ε, τα χρονικά ζητήματα που συνδέονται με αυτό για τις χώρες ΕΖΕΣ. Ε, χαίρομαι και εγώ εξ ονόματος του Σαντιάγο ε, Φίσες, ε, ε, με χαρά δηλαδή να ακούσω και εγώ όσα έχουν να πει οι συνάδελφοι, να τα σημειώσω να το, το διαβιβάσω. Ευχαριστώ πολύ. Ξέχασα να πω Ποια έκθεση είναι αυτή, να εκφωνήσω τον τίτλο. Είναι πρόταση ε, διεύρυνση της ε, πολιτιστικής σας από το 2020 στο 2030. Εισηγητής είναι ο κύριος Σαντιάγο Φίσας. Και μας είπε η Σαμπίνε Φερχάιν τα όσα σκόπευε να πει ο εισηγητής. Παρακαλώ τους και οι εισηγητές να λάβουν το λόγο. Η συνάδελφος Χιμένες Μπάρβα ζήτησε ήδη το λόγο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι στηρίζω και συγχαίρω τον κύριο Φίσας για την έκθεση αυτή. Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολύ τεχνική η έκθεση αυτή. Απλώς θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει το θέμα αυτό οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες να διευρυθούν και σε τρίτες χώρες. Πολλέ φορέ έρχονται άνθρωποι και μα πιάνουν και μα λένε: Εμεί δεν είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά αισθανόμαστε Ευρωπαίοι. Και θα πρέπει να ε, διευρυνθεί και να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια. Και επίση χαίρομαι για τι πρωτοβουλίε αυτέ, γιατί προάγεται αυτή η ιδέα η ευρωπαϊκή ότι όλοι ανήκουμε ε, στον ίδιο χώρο, στο ίδιο σπίτι, στην ίδια αιστεία και υπογραμμίζουμε ακριβώς αυτά που μας ενώνουν και ενισχύεται αυτή η, αυτό το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, Χέλγα Τρούπελ. Και εγώ θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα. Η πολύ καλή εμπειρία που είχαμε με τις πολιτικές πρωτεύουσες σε όλη την Ευρώπη καλό θα είναι να επεκταθεί και σε τρίτες χώρες. Γιατί ξέρουμε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσε ε, είναι ένα θεσμό που αφορά την επικοινωνία, την ε, ε, συμπερίληψη, δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους να συναντιούνται, να αντελάσσουν εμπειρίες, πολιτιστικά αγαθά και έτσι διευρύνεται και η δυνατότητα συμμετοχή και στο ευρύτερο κοινό. Επομένω είναι ένας πολύ καλός ρόλος να αποτελέσουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι και πρεσβευτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αυτό ο θεσμό μάλλον. Ε, νομίζω λοιπόν ότι είναι μια θετική προσέγγιση και τη στηρίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σιλβία Κώστα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι είναι μια πολύ σημαντική ιδέα αυτή που δεν είχαμε προωθήσει από την προηγούμενη θητεία. Ε, κρίμα που δεν είναι εδώ ο αρμόδιος συνάδελφος, στον οποίο θα ήθελα να πω απευθεία κάποια λόγια να τον ευχαριστήσω για το έργο του. Έτσι κι αλλιώς, ε, το Νόβισαντ είναι η πρώτη πόλη που έχει προταθεί ως ε, πρωτεύουσα αυτών των περιοχών για το 2021. Πρόκειται για μια επιτυχημένη εμπειρία που διαρκεί εδώ και μια τριακοντά ετία. Θέλουμε και την απαραίτητη στήριξη από τον προπολογισμό, διότι πραγματικά ε, η πρωτοβουλία αυτή έχει δώσει πολύ, πολύ μεγάλα ωφέλη ε, στις ε, ε, χώρες όπου εφαρμόστηκε και να πω ότι στη δική μου τη χώρα και την ε, Αγγλία έχουμε εφαρμόσει το σύστημα της πολιτιστικής πρωτεύουσας εντός της χώρας κάθε χρόνο, ετησίως. Αυτό για την πολιτιστική μας κληρονομιά και τον πολιτιστικό μας πλούτο είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να υπάρξει μια διασύνδεση και με άλλες χώρες. Ε, σε άλλε περιοχέ του κόσμου, όπω ε, μεταξύ των αραβικών πόλεων λόγω χάρη, υπάρχει αυτή η παράδοση, είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να καλλιεργηθεί ω βαλίστη στην πρακτική για το διπολιτισμικό μα διάλογο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τζούλι Και um, εγώ θα ήθελα να στηρίξω αυτή την πρόταση ο θεσμό τη Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα ήταν ένα από του θεσμού που βοήθησε και την πόλη του Λίβερπουλ στην αναγέννησή τη, ε, όταν η δυτική μα ε, κυβέρνηση αποφάσισε ότι απλώ ε, θα το αφήσουν στη δίχη του το Λίβερπουλ. Επομένω, ο πολιτισμό ήταν πραγματικά ένα θεσμό κλειδί σε ό,τι αφορά την επιτυχή μεταγενέστερη πορεία των πολεών μα. Εντάξει, έχουμε αυτή την καταστροφή με το Brexit στον Βασίλειο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε ένα, μια διέξοδο για τις πόλεις μας που τάχθηκαν περισσότερο με την παραμονή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγαλύτερη πόλη στην περιφέρειά μου είναι το Μάνσεστερ και ξέρω ότι θέλουν ε, όσο μπορούν να διατηρήσουν τους ευρωπαϊκούς δεσμούς τους. Και αυτό συντάσσεται πολύ καλά και με το Ευρωπαϊκό ε, Δίκτυο Πόλεων το οποίο και πάλι δεν αφορά μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ευρύτερο. Αυτή τη στιγμή το, το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέρμιχαμ έχει τεθεί επικεφαλής προεδρεύει δηλαδή του φορέα αυτού και ε, συνομιλώ με τους ε, συναδέλφους του Μπέρμιχαμ για αυτή τη ε, διαδικασία. Τη στερίζω πλήρως λοιπόν την διαδικασία. Ευχαριστώ κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι και η συνάδελφος Ζούντι θα το ανέφερε, αλλά πρέπει αντίστοιχα να μιλήσουμε και για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, στο πλαίσιο του θεσμού μετά τον Brexit, γιατί θα βρεθεί εν κενό, δεν θα είναι ε, υποψήφια χώρα, θα πρέπει όμως ε, κάπως να συμπεριλάβουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο, να έχουμε δυνατότητα συμμετοχή, γιατί και η βρετανική κουλτούρα είναι σημαντική για όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι λοιπόν μια νέα πρόκληση για όλου μα. Πώ γίνεται να μην αφήσουμε εκτό το Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίω όλοι ε, υποστηρίζουμε και την συμμετοχή των Βρετανικών πόλεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σολιεύσκη. Ε, Ευχαριστώ. Αρχικά θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Κάποιοι μιλήσατε για τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει ε, να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα αφορά τρίτες χώρες με την ε, ε, κοινή έννοια όπως χρησιμοποιείται στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά ε, αναφερόμαστε συγκεκριμένα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στις χώρες ΕΖΕΣ. Και για να επανέλθω σε ένα προηγούμενο σχόλιο, είναι αρκετά πιθανό το Ηνωμένο Βασίλειο να καταλήξει ακριβώς σε αυτόν τον χώρο. Για τα έτη 2020 με 2023, λοιπόν, σίγουρα θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα. Βέβαια, πρώτα θα πρέπει να υπογραφεί η συμφωνία. Κάτι άλλο που ήθελα να πω. Θα ήταν σκόπιμο αυτό το πρόγραμμα να έχει έναν προκαθορισμένο κατάλογο μελών. Υπενθυμίζω ότι και στο παρελθόν είχαμε περιπτώσεις όπου ορισμένες πόλεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν, για παράδειγμα η Κωνσταντινούπολη. Και μετά, από ό,τι θυμάμαι, αποφασίστηκε για παράδειγμα, με το Σαράγεβο, το Σαράγεβο υπέβαλε υποψηφιότητα, αλλά απερίφθη υποψηφιότητα. Τώρα μιλούμε για τις χώρες ΕΖΕΣ και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και επεκτείνουμε τον ε, θεσμό προς νέες χώρες που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση επιμέρους πολιτιστικών έργων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γεωγραφικά βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να είμαστε ακριβοδίκαιοι και να βρούμε και τη σωστή λύση. Αν ε, και δεν θα είναι μια γρήγορη διαδικασία. Και κάτι τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα είναι ένας πολύ καλός θεσμός. Από την άλλη, αν δείτε τις πόλεις μας, δεν αξιοποιούν όλες οι πολιτιστικές πρωτεύουσε ε, στο έπακρο τις ε, δυνατότητες που τους παρέχονται και ούτε είναι πάντα επιτυχή η διαδικασία. Το Λίβερπουλ, για παράδειγμα, ή το Έστεν στη Γερμανία, που έχει αλλάξει πλήρω ε, το πρόσωπό του ε, πρόσωπο της ω πόλη. Ε, και στη Βαρκελόνη, πολύ διαφορετικό, αλλά εκεί ήταν και δική του απόφαση. Υπήρξαν λοιπόν πόλει που δεν ήταν απόλυτα επιτυχείς, Όχι και απο... αποτυχίε, αλλά όχι απαραίτητα πλήρω επιτυχίες και δεν ήταν ε, πάντα ε, μακροπρόθεσμες οι αλλαγές. Ευχαριστώ. Έχω την κυρία Μπίλτ τώρα και αν δεν θέλει κανείς άλλος το λόγο, να κλείσουμε τον κατάλογο και να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Merci, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών υπάρχει από το 1985, προκειμένου να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλομορφία. Μα φαίνεται πολύ συνετό η πρωτοβουλία αυτή να υπάρχει τη στιγμή που η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά φαίνεται να απειλείται. Κυρίω ο πολιτισμό. Και σε άλλα μέρη του κόσμου όπω την Παλμύρα. Θέλετε βεβαίως να επεκταθεί και σε υποψήφιες χώρες ε, προς την, για την προσχώρηση η πρωτοβουλία αυτή. Τι θα γίνει με την Τουρκία, λόγω χάρη που είναι υποψήφια χώρα, η οποία όμω έχει πει ότι δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα και μεταξύ αυτών και στη Δημιουργική Ευρώπη. Επίση, δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτό το κοινοβούλιο μιλάμε από το 8 το βράδυ για το γεγονό ότι μα λείπουν κονδύλια για, την, για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, αλλά όλο παραδόξω προτείνεται να επιδοτηθούν ε, πόλεις και κάτι μέλη μέσα αυτής της πρωτοβουλία. Βλέπω λοιπόν να λέτε πόσα είναι τα θετικά, αλλά φαίνεται ότι πάνω απ' όλα υπερτερεί το χρήμα. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρίσταται. Θέλει να τοποθετηθεί για την έκθεση Όχι, από ό,τι φαίνεται. Η Σαμπίνε Φερχάιν, εκπροσωπώντας τον Σαντιάκο Φίσα, θες να πεις τίποτα άλλο, να προσθέσεις τίποτα. Εξ ονόματος του Σαντιάγο Φίσας θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και να ξεκαθαρίσω το εξής, για να μην το αφήσω αναπάντητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει λεφτά για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες ε, χωρών που δεν ανήκουν σε αυτή από τον Ευρωπαϊκό Κόρβανα. Τα κράτη που συμμετέχουν ε, συνεισφέρουν, έχουν ένα ποσοστό και συμμετέχουν στη χρηματοδότηση. Και καλά κάνουν. Δηλαδή, αν συμμετέχουν ενεργά, θα πρέπει να παίρνουν το μερίδιο που του αναλογεί από τον προπολογισμό. Δεν παίρνουν έτσι λεφτά από την Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Όντω ισχύει αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν η Τουρκία στο μέλλον αποφασίσει να αποσυρθεί από το πρόγραμμα αυτό, δεν πρόκειται να χρηματοδοτούνται και τα έργα από το πρόγραμμα Creative Europe της Δημιουργική Ευρώπη. Αυτά είναι σαφή και ξεκάθαρα και ρυθμισμένα. Και κατά τα άλλα το κύριο βάρος των πολιτιστικών πρωτεύουσων το φέρουν οι ίδιες οι πρωτεύουσες. Και τακτικά. Όχι μόνο απαιτείται κάτι τέτοιο, αλλά το αναλαμβάνουν το κόστος αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Πρέπει να σας πω επίσης ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών έχει οριστεί 30 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, την άλλη Δευτέρα. Η δε ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μας θα διεξαθέσει 28 Φεβρουαρίου. Επόμενο θέμα, αριθμών 7. Συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ε, ανταγωνιστικότητα και συνοχή. Η ευρωπαϊκή κοινωνία ε, Gigabyte και 5G. Η συγκίτρια είναι εδώ η κυρία Σίλβια Κώστα. Έχουμε σχέδιο γνωμοδότησης εμείς να συζητήσουμε τώρα και να εξετάσουμε και αμέσω το λόγο στην κυρία Σιλβία Κώστα. Ένα τρίλεπτο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως τα είδατε, από το σχέδιο έκθεσης, όπου υπάρχει περιορισμό στους χαρακτήρες, δεν μπορούσα να περάσω σε όλες τις λεπτομέρειες όσο θα ήθελα. Προσπαθούμε να παρουσιάσουμε την ε, όλη αυτή κοινωνία των gigabyte και της τεχνολογίας των, του 5G ως μια ευκαιρία για τα οπτικοακουστικά, για όλη τη δημιουργική βιομηχανία, για την πολιτιστική μας κοινωνία. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική έχει το φιλοδόξο στόχο μέχρι το 2025 να έχει υπερταχή ίντερνετ και να το προσφέρει σε όλους, ακόμα και στα δημοτικά και δευτεροβάθμια σχολεία και βιβλιοθήκες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα και ελπίζω με περαιτέρω τροπολογίες να επεκτείνουμε αυτό το στόχο και στα πανεπιστήμια. Η πρόκληση είναι μεγάλη και για τις εκπαιδευτικές μεθόδους. Μιλώ για το e-learning και το e-teaching για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και ούτω καθεξής. Πρόκειται λοιπόν για μια θετική εξέλιξη, η οποία σχετίζεται άμεσα με τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι και τις εκπαιδευτικές μας προκλήσεις. Κάτι άλλο που βρίσκω σημαντικό είναι να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα. Γίνεται και αυτό θεμελιώδου σημασία, καθώς και η λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το πώς επηρεάζουν τον πληθυσμό διότι η ψηφιακή διάσταση της ιδιότητας του πολίτη παίρνει μεγαλύτερη σημασία. Ταυτόχρονα, η διάδοση του 5G μπορεί να δώσει και άλλες ευκαιρίες με νέα περιεχόμενα πολιτιστικά και δημιουργικά online και με την διαδραστική παράμετρο σε λειτουργία. Δηλαδή μπορεί κανείς να είναι ταυτόχρονα δημιουργός και ε, ε, ε, τέκτης των ερεθισμάτων αυτών. Με την αλυσίδα όλων των αξιών των οπτικοακουστικών μέσων να ενισχύεται. Ακόμη μια υπογράμμιση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει ακόμη περισσότερο υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εκπομπής στο ραδιοφάσμα Και γι' αυτό προαναγγέλλω ότι επί του σημείου αυτού θα ακούσω βέβαια τις απόψεις των υπολείπων, αλλά θα είμαι λίγο πιο αυστηρή στον ορισμό. Με μια πιο συγκεκριμένη παράγραφο εδώ. Είναι ένα από τα θέματα για τα οποία πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Κάτι άλλο που δεν μπόρεσα να καλύψω εδώ λόγω του περιορισμού στην έκταση της έκθεσης είναι η ασφάλεια του δικτύου. Δεν αμφιβάλλω ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ διότι όσο περισσότερο υπάρχει διάδοση τη τεχνολογία, ακόμη και με το διαδίκτυο των πραγμάτων, των, των πραγμάτων, γίνεται τόσο ατελείωτο το φάσμα των προϊόντων και των φορέων που δρούν σε αυτό το διαδίκτυο και των πληροφοριών που διατίθενται. Οπότε πρέπει όλο αυτό να συμβαδίζει με τη βεβαιότητα ότι υπάρχει επαρκής παροχή προστασίας η network security όπως θα μπορούσαμε να την πούμε. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίζουμε αυτήν την προστασία των πληροφοριών και του λογισμικού. Εκεί νομίζω που να εμβαθύνουμε περαιτέρω και επιπλέον χρήσιμο θα ήταν να δώσουμε έμφαση στο σημείο που αφορά τι διαφορέ μεταξύ μελών. Ήδη το τονίσαμε σε σχέση με την έκθεση περί ραδιοφάσματο, το τι διαφορέ υπάρχουν μεταξύ των μελών στη δυνατότητα διασύνδεση με το υψηλή ταχύτητα ίντερνετ. Πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη, ώστε η τεχνολογία 5G να μην μεγαλώσει κι άλλο αυτό το χάσμα, αλλά να υπάρξει αρμονική ανάπτυξη όλων των 100 μελών προ την ίδια κατεύθυνση. Όχι να ενταθούν οι διαφορές. Ευχαριστώ και περιμένω τις αντιπράξεις των σχεδόν. Ευχαριστώ πολύ, Σίλβια. Η Σαμπίνα Φεχάιν. Χαίρομαι που ως Επιτροπή Πολιτισμού έχουμε λόγο για αυτό το θέμα και γνωμοδοτούμε. Γιατί είπε ορισμένα στοιχεία η Σίλβια Κώστα που μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν η τεχνολογία κινητών της πέμπτης γενεάς δεν έχει να κάνει μόνο με το γρήγορο ίντερνετ. Αυτό μπορείς να το βρεις και από αλλού. Αλλά αυτό το 5G αφορά τα κινητά τηλέφωνα ε, και έχει και πολλά στοιχεία και πτυχές που αφορούν τον πολιτισμό, τη δημιουργία, πολλά πράγματα που παράγονται και καλό είναι να γνωμοδοτούμε κι εμείς. Προσοχή όμως, ε, όσο διευρύνεται αυτή η τηλεφωνία πέμπτης γενεάς και τώρα που το είπες, το πρόσεξα και εγώ, γιατί λείπει από το κείμενο, θα πρέπει να φροντίσουμε άλλες ε, μορφές ε, μετάδοσης να μην χαθούν όπως, ε, ή να μην περιοριστούν, όπως είναι οι ραδιοσυχνότητες όπου εκπέμπουν τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Δηλαδή να μην τα διζώσουμε όλες τις συχνότητες στην τηλεφωνία, να υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης και εκεί. Το δίκτυο 5G είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ιδιαίτερα ε, ε, για να ξεπεραστεί το ψηφιακό χάσμα και αυτή η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην Ήπεθρο και τις αστικές περιοχές. Γιατί αν έχουμε ευρυζωνικότητα, αυτή σήμερα την έχουμε στις πόλεις και εκεί δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα γιατί εκεί παράγεται και η οικονομία και αξίζει και μάλλον αποφέρει ε, η ευρυζωνικότητα, ενώ στην Ήπεθρο δεν συμφέρει τόσο πολύ ε, να δημιουργείται αυτή η υποδομή. Ε, δεν συμφέρει να επεκταθεί το δίκτυο για σταθερά τηλέφωνα συσκευές και υπολογιστές, όχι όλα μέσω της κινητής τηλεφωνίας λοιπόν. Σίγουρα θα μπορέσουμε να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες ε, τι γίνεται με την ε, παιδεία. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ε, ποιες είναι ευκαιρίες που δημιουργούνται με το γρήγορο διαδίκτυο και στα κινητά. Έχουμε νέους τρόπους εξωσχολικής εκμάθησης ή εξω διδασκαλική, δηλαδή εκτός της αίθουσας διδασκαλίας μπορεί κανείς να ε, συνδυάζει πολύ ωραία πράγματα που δεν ε, έχουν να κάνουν με το σχολείο αυτό καθ' αυτό και την αίθουσα ε, όπου θα γίνεται το μάθημα. Μπορεί να γίνεται το μάθημα αλλού με πολύ ωραίους τρόπους και με πολλές ευκαιρίες. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Thank you, and welcome to your... Ευχαριστώ και συγχαρητήρια την άλυψη των καθηκόντων σα. Η συνάδελφο Μακλάρκιν δεν ήταν, μπορούσε να έρθει εδώ σήμερα ε, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Όμω ε, μου, μίλησε, μου ζήτησε να μιλήσω ο ονοματό τη και χαίρομαι ιδιαίτερω γιατί είμαι εισηγητή, όχι σκιώδη ε, για μια φορά, στην Επιτροπή Ρέτζι για αυτό το φάκελο. Μου ζήτησε λοιπόν να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει για αυτή την ομοδότηση μέχρι σήμερα. Γενικά οι Ευρωπαίοι στρατηγικοί μεταρρυθμιστέ ε, στηρίζουν ε, την πρόταση και υπάρχει ευρύτερη στήριξη σχετικά με την πρόταση αυτή σε όλο το Κοινοβούλιο, παρότι υπάρχουν προτάσει διαφορετικέ. Ο σκοπό λοιπόν τη κοινωνία αυτή είναι πολύ γνωστό και φιλόδοξο. Απαιτεί λοιπόν μία ε, μελλοντοστράφη προσέγγιση και έγκαιρη αντίδραση σε ό,τι αφορά τις αλλαγές ε, στην κοινωνία μας. Είναι τεράστια η κλίμακα των ε, αλλαγών και οι προκλήσεις για τους επενδυτές και για τους παρόχους υπηρεσιών. Και η υψηλή ποιότητα συνδεσιμότητα είναι πολύ σημαντική και για τον Βασίλειο και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε αύξηση αριθμού των παρόχων που δίνουν λοιπόν τέτοιες ε, υπηρεσίες ε, καλής ποιότητας και καλού περιεχομένου και δημιουργούν και θέσεις εργασίας. Ιδίω σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει τώρα, θα πρέπει να έχουν τη θέση, ε, τη δυνατότητα να ανταγωνίζουν τι μεγαλύτερε σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να του δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία και καθήκοντα. Δεν θα πρέπει λοιπόν οι οι δικοί μας ε, φορείς και πάροχοι να ε, μείνουν πίσω σε σχέση με τους ε, Αμερικανούς που έχουν προχωρήσει τεχνολογικά σε μεγάλο βαθμό, ήδη έχουν περάσει δηλαδή στην τεχνολογία 5G. Αυτή λοιπόν η συνδεσιμότητα μπορεί να ενθαρρύνει και την επιχειρηματικότητα, αλλά και για να περιορίσει τα γραφειοκρατικά άχθη και να διευκολύνει τι υπηρεσίε κατάρτιση, για παράδειγμα, όπω αναφέρθηκε προηγουμένω. Αναγνωρίζουμε λοιπόν την, και χαιρετίζουμε την αναγνώριση δυνατοτήτων για την κατάρτιση και ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί την προσπάθεια, καθώ και η ανταλλαγή των πρακτικών. Βέβαια, αυτή η φιλοδοξία δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για περιττή ρύθμιση και ρυθμιστικό πλαίσιο. Όταν αυτό μπορεί λοιπόν να τύχει ρύθμιση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να το επιτρέπουμε. Για παράδειγμα, ενώ προτείνει 25 ετή άδειε η πρόταση για τι άδειε λοιπόν ραδιοφάσματο και αυτό μπορεί να ε, δημιουργήσει προβλήματα για τι επενδύσει, θα πρέπει να υπάρξουν, ε, να ζητήσουμε στοιχεία που να δικαιολογούν την περαιτέρω κεντροποίηση και συγκέντρωση μάλλον τη πολιτική και τέλος, ε, θέλουμε το 5G για να δίνουμε μεγαλύτερη ε, πρόσβαση σε περιεχόμενο υψηλού επίπεδου, όμω θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τη διάσταση των ε, δικαιωμάτων γενοτικής ιδιοκτησία, ούτω ώστε το 5G να μην επιτρέπει, απλώς να μην διευκολύνει την παράνομη λήψη ιδιωτικού περιεχομένου και θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά και το τι ακριβώς ε, είναι το 5G, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφής ο ορισμός, παρότι χρησιμοποιείται δεξιά και αριστερά αυτός ο όρος. Τι είναι όμως τελικά, τι θα γίνει, τι θα αποτελέσει όταν έρθει. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου, γιατί νομίζω ότι ο ορισμός του 5G είναι ε, πολύ πιο ασαφή σε σχέση με τον ορισμό του 4G και 3G όταν ε, είχαν προκύψει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρευρίσκεται. Θέλει να λάβει και το λόγο. Uh, yet because the... Όχι ακόμα δεν έχει έρθει ακόμα εμπειρογνώμονα, γιατί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα ε, προβλεπόταν για τι 4.30. Έρχεται λοιπόν η εμπειρογνώμονα μα. Μπορούμε να καταγράψουμε τι ερωτήσει σα και όταν έρθει να απαντήσει. Good. Ε, καλώς. Κρίμα που απουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Σίλβια Κώστα για να κλείσει. Για να πω προηγουμένως όμως η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών είναι 30 Ιανουαρίου στις 4 το απόγευμα την άλλη Δευτέρα η δε ψηφοφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται για τις 22 Μαρτίου. Σίλβια. Να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδες συναδελφούς ε, όπως έκανα και στην αρχή, να πω ότι η αναφορά σε θέματα που αφορούν την επέκταση του 5G και το τι γίνεται με τα blockbuster σε σχέση με αυτήν την ε, ανάγκη είναι κάτι που το έχω υπόψη. Ε, τα είπα λίγο συνοπτικά βέβαια, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ίσως με μια τοπολογία. Και αυτό που υπόθηκε για το copyright, συμφωνώ και έπειτα. Χρήσιμο νομίζω θα είναι να εξετάσουμε όλο το φάσμα των θεμάτων όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, ίσως μπαίνοντα και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαι πολύ ανοιχτή στις προτάσεις σας. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει ορισμός του ραδιοφάσματος, όπως έγινε και με την ψηφιακή στρατηγική, είναι ένας ορίζοντας απαραίτητος εντός τόπου που να ενταχθούν όλα τα υπόλοιπα, αναγνωρίζοντας τις ε, ιδιαιτερότητες των διαφορών χωρών και τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες όλα αυτά μπορούν ε, να προχωρήσουν. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα με τα Block Blaster, την παιδεία και όλα αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να πω ότι τα ωράρια στην ημερήσια διάταξη είναι ενδεικτικά και ε, έτσι, χονδρικά. Και επειδή ε, είχαμε εκλογές, καμιά φορά χρειάζεται να υπολογίσει κανείς ότι μήπως χρειαστεί μυστική ψηφοφορία. Γι' αυτό ήταν αυτό το ωράριο και δυστυχώς, ε, ευτυχώς δεν ξέρω, τελειώσαμε πάρα πολύ νωρίτερα εξού και διαβεβάστε στη συνάδελφο ότι δεν χρειάζεται να έρθει πια οι σκιώδεις και οι αν χρειαστεί κάτι θα αποτανθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. απλώ να ξέρουμε ότι είναι ενδεικτικά τα ωράρια που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Και αν χρειαστεί λοιπόν θα το ρολίσουν διμερό. Ευχαριστώ πολύ Σίλβια, ευχαριστώ πολύ και ε, όσους έλαβαν το λόγο. 30 Ιανουαρίου στις 4 το απόγευμα λίγη προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Συνεχίζουμε. Ε, εδώ ολοκληρώνεται το δημόσιο τμήμα ε, της σημερινής μας συνεδρίασης και θα παρακαλούσα όλους εκείνους που δεν είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που δεν εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποχωρήσουν, διότι έχουμε και ένα σημείο και κλεισμένων των θυρών. Και πρόκειται για ένα θέμα τριμερούς διαλόγου. Και αυτά μας αρέσει να τα συζητάμε μεταξύ μας. Αύριο το πρωί, 9 η ώρα, συνεχίζουμε τη δημόσια συνεδρίαση. Παρακαλώ να είστε όλοι στην ώρα σας για να αρχίσουμε ψηφοφορίες 9 η ώρα ακριβώς. Έχουμε 6 ψηφοφορίες στην ημερήσια διάταξη και κατά τα άλλα πολύ σφιχτό και βαρύ πρόγραμμα. Έχουμε τις πραγματικές δηλώσεις της Μαλτεζικής Προεδρίας και άλλα θέματα πολλά. Οπότε, αν αργήσουμε να αρχίσουμε θα έχουμε λιγότερο χρόνο για τη συζήτηση. Θα παρακαλούσα λοιπόν να αρχίσουμε στην ώρα μας για να προχωρήσουμε και να έχουμε χρόνο για συζήτηση κανονική το πρωί. Αυτά. Αποχώρησαν όλοι οι εξωτερικοί. Mm. Περιμένουμε ένα λεπτάκι ακόμα.